Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η... επαναλαμβάνεται η συνεδρίασή μας. Τα συνοπτικά ε, πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης έχουν διανεμηθεί. Υπάρχουν παρατηρήσεις. Δεν βλέπω να υπάρχει αντίδραση στην αίθουσα, οπότε θεωρούμε ότι τα πρακτικά εγκρίνονται. Τώρα ερχόμαστε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, που είναι δηλώσει...